Το κείμενο αυτό θα το βρείτε στην, ε, στον ιστότοπο Seance en Direct και με αυτόν τον τίτλο στα πρακτικά θα δημοσιευτεί την ε, Τετάρτη σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού με τον πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψω πέντε νομοθετικές πράξεις ε, που εγκρίθηκαν ως αφορά νομοθετική διαδικασία. Τα κείμενα αυτών των πράξεων θα δημοσιευθούν στα πρακτικά τη σημερινή μα συνεδρίασης. Αγαπητοί συνάδελφοι, την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε την ε, Παγκόσμια ημέρα γυναικών. Η ισότητα γυναικών και ανδρών είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες